Okay, welcome to this meeting. Χαίρετε. Υπάρχουν θέσεις πίσω. Καθίστε παρακαλώ. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση αυτή. Τώρα θα αρχίσω τα σουηδικά. Άμα δεν γνωρίζετε σουηδικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας. Den eh, eh, Χαίρετε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι, τότε λέω να τα εγκρίνουμε, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Τρία. Ανακοινώσεις του Προέδρου ή της Προεδρίας. Δεν υπάρχουν για σήμερα πάει και αυτό. Μια στιγμή παρακαλώ μου διαφεύγει. Punkten 4 är eh, justering av protokoll. 4. Έγκριση των πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων. Αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκριθέντα. 5. Πέντε. υπάρχει εδώ μια αλλαγή, μια αλλαγή, δεν είχα την ίδια ημερήσια διάταξη, γι' αυτό, γι αυτό μου είχε διαφύγει. Λοιπόν, το 5 επαναλαμβάνω, ανακοινώσει του Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών και συντονιστριών. Νομίζω κάτι έχετε στους φακέλους σας για αυτό το θέμα. Αν δεν ακούστούν πάλι αντιρρήσεις και αυτό που έχετε στους φακέλους σας εγκρίνεται. Και τώρα θα χορηγήσω την Προεδρία εδώ στη συνάδελφο. Good Χαίρετε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που θα προεδρεύσω στις ψηφοφορίες, στην σημαντικότατη αυτή ψηφοφορία που γίνεται για δεύτερη φορά για μένα. Καθόλα τα έτη της εργασίας μου εδώ. Η έκθεση αυτή είναι της Εύας Μπριτ Σβένσον της προηγούμενης Προέδρου αρχίζει. Είναι όλοι και όλες έτοιμοι. Τροπολογία 4. τέσσερα Α, με συγχωρείτε. Πρώτα ο πρόεδρος. Ναι, λοιπόν, άλλαξα θέση και ρόλο. Όπως είπε η πρόεδρος η Εύα Μπριτ Βένσον είχε γράψει την έκθεση αυτή και χαίρομαι που φτάσαμε στο τέρμα αυτής της διαδικασίας γιατί με ενδιαφέρουν και μένα πολύ τα θέματα ισότητας, πάρα πολύ. Και η βασική μέθοδος που επέλεξε η συγκήτρια είναι νομίζω σωστή. Πιστεύω ότι η προοπτική της έχει πολύ μεγάλο μέλλον και πρέπει να την αναφέρουμε παντού και πάντοτε. Υπάρχουν μερικές τροπολογίες που κατατέθηκαν, όχι πάρα πολλές. Και νομίζω ότι όλες εκτός από δύο είναι αποδεκτές. Γίνονται αποδεκτές. Εγώ μπορώ να τις δεχτώ δηλαδή. Ιδίω την 3 και 6 και 7. Και 7. 7. Ναι, ναι, αυτές που δεν δέχομαι είναι οι 4 και 5. Δεν σας τις συνιστώ αυτές. Γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των φίλων εδώ στη μεταχείρισή τους δηλαδή. Αυτό είναι νομίζω κάτι που δεν το δέχεται πια κανείς. Και μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα στη μεταχείριση των δύο φίλων. 50-50%. Σας ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 4 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο ηλεκτρονικά. Μάλιστα έχετε όλες τις κάρτες σας τότε. Εντάξει. Λοιπόν, αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α, δεν είναι έτοιμο το μηχάνημα. Μια στιγμή να ετοιμαστεί. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 12-8 ή 8-12. Ορίστε κυρία Μπάστος. χωρίς μικρόφωνο. Α, τότε καλά. Αν θέλετε μπορούμε να ψηφίσουμε με πολλές, πολλές τροπολογίες μαζί. Όχι. Α, εντάξει, όχι. Λοιπόν, έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επτά υπέρ. Κατά εποχές Επαλήθευση για την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχισε. Ωραία. 13 υπέρ, 11 κατά, μία, καμία αποχή εγκρίνεται. 8. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κυρία Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι αν είναι αποδεκτή η 9. Γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε ειδική μεταχείριση για την Επιτροπή Γυναικών σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις επιτροπές, για όλες τις επιτροπές και νομίζω ότι δεν είναι αποδεκτή αυτή η τροπολογία. Α, τότε καλά. το καλύτερα. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ για αυτό που είπατε, αλλά εδώ μιλάμε για την Επιτροπή ΑΦΚΟ που είναι η αρμόδια και εκείνη μπορεί να την δηλώσει αποδεκτή ημί. Ναι, αλλά τέτοιου είδους διαδικασία πρέπει να αναλυθεί για όλες τις επιτροπές δεν μπορούμε να ζητάμε κάτι ιδιαίτερο για την Επιτροπή Γυναικών που να μην ισχύει για τις άλλες επιτροπές. Αυτό λέω. Καλά. Θα το δούμε. Ας το αφήσουμε για την Ολομέλεια. Ψηφίζουμε τώρα και θα κρίνει η Ολομέλεια. Εν τω μεταξύ η γραμματεία θα ελέγξει.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 για την 14. Ένας σοσιαλιστής παραπάνω βρέθηκε. Ξανάρχεται η ψηφοφορία. Ξαναρχίζει. Έληξε. 13 κατά απορρίπτεται 15 υπέρ κατά απο, εγκρίνεται α καλά επαλήθευση επαλήθευση για την 15 άρχεται η ψηφοφορία έληξε εγκρίνεται ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική και συνολική ψηφοφορία για το κείμενο έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλεξε. Εγκρίνεται 24. Συγχαρητήρια.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 Okej, då Συνεχίζουμε. Το 7. Προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία στον ορίζοντα το 2020. Η κυρία Μπος Κιούρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, η την τελευταία έκθεση που έκανα για την κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία, η τελευταία μου έκθεση έγινε το 2007. Καιρός ήταν λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Η κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία χειροτέρευε από ό,τι διάβαζα από τον τύπο αν κρίνω από τις δολοφονίες γυναικών ερεύνησα, οργάνωσα ακρόαση και πήγα δύο φορές στην Τουρκία για να δω τα πράγματα όμως Μίλησα με πολλούς ενδιαφορόμενους, 7 υπουργού, μεταξύ των οποίων τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον Υπουργό Οικογενειακών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Εργασίας, Παιδείας και Οικονομικών. Μίλησα και με πολλούς κοινοβουλευτικούς και από κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς και με προσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις γυναίκες. Μίλησα και με τα συνδικάτα. Ε, επισκέφθηκα διάφορα άσυλα γυναικών θυμάτων βίας και μίλησα και με γυναίκες από διάφορους οικονομικούς τομείς και περιφέρειες. Το θέμα της βίας κατά των γυναικών του χαμηλού μορφωτικού τους επίπεδου και της χαμηλής τους ειδίκευσης. Τα είδα όλα αυτά και τα ανέφερα στην έκθεσή μου καθώς και συστάσεις για βελτιώσεις. Αλλά επίσης είδα και θετικές εξελίξεις. Έχει σχεδόν κλείσει το χάσμα στη, μεταξύ των δύο γενών στην παιδεία στο εξή θα θεωρείται υποχρεωτική εκπαίδευση στην Τουρκία για όλα και για τα δύο φύλλα και έχουν ληφθεί αυστηρότερα μέτρα για και κυρώσεις κατά των εγκλημάτων και της βίας κατά των γυναικών και υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων ως προς αυτό το θέμα. Στην έκθεσή μου κάνω και μερικές συστάσεις ιδιαίτερα στον τομέα της βίας κατά των γυναικών, των γυναικείων ασύλων και κέντρων περίθαλψης, το θέμα της μερικής απασχόλησής τους και ιδιαίτερα ζητάω μηδενική ανοχή για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Στο παρελθόν η Τουρκία είχε δεχτεί τέτοια μέτρα για τα βασανιστήρια και τα αποτελέσματα ήταν αρκετά θετικά. Ονόμασα την έκθεσή μου μια προοπτική στον ορίζοντα του 2020 και θεωρώ ότι μία προτεραιότητα του ορίζοντα αυτού είναι μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή. Σε όλες μου τις ε, συνεννοήσεις και συνεντεύξεις και τις επαφές μου κατάλαβα ότι κάτι το κοινό υπήρχε με όλα τα προβλήματα μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολιτευμένων κομμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ώστε οι πατριαρχικές δομές της κοινωνίας να βασίζονται στο εξή στην ισότητα των φύλων. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να πάψει η βία κατά των γυναικών και να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην εξουσία και την εργασία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, γιατί μια τέτοια αλλαγή θα πραγματοποιούνταν καλύτερα μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού δημιουργίας προτύπων για το ρόλο των γυναικών που μπορούν να ακολουθήσουν τα κορίτσια. Και δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αλλάξει η νοοτροπία. Αυτό μπορεί να ε, αποτελεί μια καμπάνια για την ισότητα των γυναικών αλλά έχει ξαναγίνει, αλλά αυτή τη φορά να συμμετάσχουν και άντρες και γυναίκες στην καμπάνια στην Τουρκία. Αυτό ήθελα να πω για την έκθεσή μου. Προσβλέπω στις αντιδράσεις σας και φυσικά σε συνεργασία γενικότερα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Όποιος θέλει το λόγο. Ποιος? Εσείς κυρία μου δεν λέω το όνομά σας για να μην το προφέρω άσχημα. Ναι, πρόεδρε, εντάξει, δεν πειράζει που δεν το λέτε το όνομά μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε ότι η κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία έχει ε, βελτιωθεί βέβαια αρκετά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο ε, ποσοστό βίας εναντίον των γυναικών. Ε, υπάρχουν πολλά που πρέπει να αλλάξουν στην τουρκική κοινωνία, πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες και αυτό ξέρω ότι κρατάει, παίρνει πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να υπάρξουν αυστηρότερες ποινές όσων ασκούν βία κατά των γυναικών και θα ήθελα ίσως να σας αναφέρω και μια περίπτωση όπου ε, υπήρξε έτσι ε, μεγάλη πρόοδος. Ε, δολοφονήθηκε 18χρονη κοπέλα από τον αδερφό της γιατί παντρεύτηκε χωρίς να ζητήσει την άδεια του πατέρα της. Όταν διαλύθηκε ο γάμος, η κοπέλα γύρισε στο σπίτι της. Ε, όλη η οικογένεια λοιπόν καθόταν στο σαλόνι και ο αδερφός της στο διπλανό δωμάτιο τη δολοφονούσε. Η αστυνομία μόνο τον αδερφό της ουσιαστικά συνέλαβε για τη δολοφονία αυτή τιμής. Νομίζω ότι κανονικά έπρεπε να συλλαβεί και όλη την οικογένεια ε, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια επανάσταση απέναντι στην αντιμετώπιση της ε, βίας. Γιατί συνήθω αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα εγκλήματα τιμή δεν θέλουν να τα κάνουν, αλλά δέχονται τέτοια πίεση από την οικογένεια για να καθαρίσουν την τιμή τη που αναγκάζονται να το κάνουν. Νομίζω λοιπόν ότι και η οικογένεια θα πρέπει να τιμωρείται ω ηθική αυτούργο. Πρέπει λοιπόν ε, να δράσουμε σε πολλά επίπεδα. Επίση, σε πολλά σημεία ε, ζητούμε από την Τουρκία να αντιμετωπίσει το θέμα της ε, βίας κατά των γυναικών και να τις προστατεύσει επαρκώς. Υπάρχουν, ε, υπάρχει και νομοθεσία βέβαια στην Τουρκία η οποία έχει αλλάξει ως προς αυτό και είναι σημαντικό να σταματήσουν αυτές οι περιπτώσεις ε, υποχρεωτικών ε, γάμων. Πρέπει οι γυναίκες στην Τουρκία να μπορούν να επιλέξουν μόνες τους τον σύζυγό τους. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή καταπίεσης. Αυτό, συνήθως αυτοί οι γάμοι γίνονται κάτω από τεράστια πίεση. Τώρα, η εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να πάνε όλο και περισσότερα κορίτσια στο σχολείο, να αντιμετωπιστεί ο αναλφαβητισμός, πρέπει να υπάρξουν ενημερωτικές εκστρατείες, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για να, αντι... να αντιμετωπιστούν του αναλφαβητισμού και οι γυναίκες να μπορούν να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί μέσα στην κοινωνία. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας γιατί μπορεί να επηρεάσει και την, το ρόλο της γυναίκας στην αγορά εργασίας που επίσης πρέπει να ενισχυθεί οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να απασχολούνται. Θα πρέπει να μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσω της καλύτερης εκπαίδευσής τους. Ας πούμε υπάρχουν τα προγράμματα μικρών δανείων που έχουν βοηθήσει να ενισχυθεί η θέση των γυναικών. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από τη Γερμανία, όπου υπάρχουν ε, πολλοί Τούρκοι τρίτης γενιάς πια. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε μετανάστες Τούρκους. Και πρέπει να πω ότι πολλοί, ε, πολλοί Τούρκοι έχουν ε, ε, αλλάξει η νοοτροπία και σκέφτονται όπως ε, εμείς. Ε, και βεβαίως υπάρχουν και στη Γερμανία περιπτώσεις οικογενειών που έχουν τη δική τους νοοτροπία, τη δική τους αντίληψη για τη θέση της γυναίκας, των δικαιωμάτων της γυναίκας. Και στη Γερμανία υπάρχουν συνέχεια τέτοιες, τέτοια άρθρα στις εφημερίδες για εγκλήματα τιμής δεν είναι εγκλήματα τιμή, είναι δολοφονίε. και είναι πραγματικά απαράδεκτο γιατί γίνονται μέσα στην, στους κόλπους της, ε, των οικογενειών. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι περιπτώσεις, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ε, ριζωμένο στην αντίληψη των ανθρώπων αυτών ότι αυτό δικαιούνται να το κάνουν ή μπορούν να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα τιμής. Πρέπει λοιπόν στις μεγάλες, πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας σαφής τρόπος αντιμετώπισης. Θα μπορούσαμε εμείς ίσως να δημιουργεί, να θέλουμε ας πούμε να έχουμε ένα νέο ε, κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο όμως θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι γυναίκες ανθρώπινα όντα είναι και έχουν δικαιώματα. Τώρα για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, που έχουμε με την Τουρκία, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να, ε, θέσουμε τις, να κάνουμε τις περισσότερες προσπάθειες. Να πούμε ότι ναι, μπορείτε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όμως σέβεστε τα δικαιώματα της γυναίκας και αν μπορείτε νομικά να την προστατεύσετε όταν, ας πούμε, την χάνει η διακριτική μεταχείριση. Πρέπει να φροντίσετε ώστε οι κόρε των γυναικών αυτών να μπορούν να πάνε στο σχολείο, Πρέπει να υπάρχει λοιπόν να υπάρξει αλλαγή νοοτροπία. να, και από εμά ε, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σταθεροί στην απόψή μα, γιατί πρέπει και η Τουρκία να κάνει κάποια πρόοδο σε αυτό. Και να πω κι άλλο ένα. Ε, υπάρχουν διάφορα προγράμματα στην Τουρκία τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, τουρκική κυβέρνηση όμως έχει μικρό ρόλο στη χρηματοδότηση, οπότε θα πρέπει και εκεί κάτι να γίνει. Εμείς επενδύουμε σε αυτά τα προγράμματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στην, στην Τουρκία, αλλά θα πρέπει και η τουρκική κυβέρνηση να κάνει ό,τι της αναλογεί. Η κυρία Μποσκούρτ όντω έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, πήγε στην Τουρκία, είδε πώ έχει κατάσταση, πραγματικά είναι μεγάλη η προσπάθεια που έκανε για την ε, γνωμοδότησή τη μπορώ να συμφωνήσω με πάρα πολλά στοιχεία. Πρέπει όντω να αναλάβουμε δράση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη θέση τη ε, γυναίκα στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Παπαδοπούλου έχει το λόγο. Sorry. Thank you very much, uh, Chair. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα προσεκτικά την έκθεση. Είναι νομίζω μια πολύ καλή προσπάθεια αυτή που κάνει η κυρία Μποσκούρτ για να καταγράψει ποιες είναι οι αλλαγές που γίνονται τώρα στην Τουρκία σε ό,τι αφορά το νόμο. Έτσι ώστε να δούμε και μέσω της Επιτροπής Ισότητας πώς έχει βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ παρακολουθώ το θέμα αυτό και των ε, υποχρεωτικών γάμων και των εγκλημάτων ε, τιμής ε, τα τελευταία 20 χρόνια μπορώ να σας πω. Ήμουνα και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχω διαβάσει και την έκθεση της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία παρά την αισιόδοξη προσέγγιση της εισηγήτριας θα πρέπει να τονιστούν γιατί δεν είναι απλό να υπάρχουν ε, κανόνες ή ε, μια σωστή νομοθεσία. Το σημαντικό είναι η εφαρμογή όλων αυτών των κανόνων και των νόμων. Η εφαρμογή δεν είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει από τις τουρκικές αρχές. Για τα εγκλήματα τιμής ε, υπάρχουν, εξεκολουθούν να είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά. Υπάρχει μεγάλη βία, μεγάλο ποσοστό βίας κατά των γυναικών, υποχρεωτική γάμη γυναικών, κοριτσιών μεταξύ 14 και 16 χρονών. Επίσης είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Επίσης το θέμα των απαγωγών είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Ο αναλφαβητισμός των γυναικών είναι πολύ ψηλά, ειδικά για γυναίκες κουρδικής καταγωγής. Είναι γεγονός, συμβαίνει, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί. Η φτώχεια επίση των γυναικών είναι σημαντική. Εγώ έχω ε, επισκεφθεί πολλέ φορέ ε, την Τουρκία ω ε, μέλο τη της, της Μικρή Κοινοβουλευτική Επιτροπή μεταξύ Ευρώπη και Τουρκία και το έχω ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Έχω ακούσει τι λένε οι γυναίκε οι ίδιε και τι λένε οι γυναίκες με κουρδικής καταγωγής για την κατάσταση αυτή. Και πραγματικά με όλο το σεβασμό το θέμα δεν είναι να συναντούμε μόνο ε, αξιωματούχους και υπουργού. Πρέπει να ακούμε και τον, τον απλό κόσμο, να ακούσουμε τη φωνή του, τη φωνή των γυναικών. Και σε ό,τι αφορά την καλύτερη, τις περισσότερες ευκαιρίες για καλύτερη εκπαίδευση, ναι, ακούσαμε ότι υπάρχουν ε, υπάρχει βελτίωση σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση τι γίνεται. Γυναίκε που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, πόσε είναι τι επαγγέλματα τελικά κάνουν, τι δουλειά βρίσκουν μετά το πανεπιστήμιο. Και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ασύλων δεν είμαι α, ικανοποιημένη, γιατί σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να υπάρχει για κάθε 50.000 ανθρώπους ένα άσυλο. Ο αριθμό των ασύλων στην Τουρκία είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν εκεί. Οπότε θα πρέπει να καταγράψουμε πολύ καλύτερα την κατάσταση εγώ θα υποβάλω πολλές τροπολογίες γιατί έχω, και, έχω υπόψη μου και την έκθεση της κυρίας Όμεν ε, πέρσι αλλά και, το, και την έκθεση τη σχετική του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εδώ στην έκθεση λέμε για το, μιλούμε για το κεφάλαιο 23. Εγώ είμαι κατά του ανοίγματο του κεφαλαίου 23 και θα σα πω γιατί. Είναι πολιτικό το θέμα. Θα ξέρετε ότι το Συμβούλιο ε, μιλά για, την, για το άνοιγμα των 8 κεφαλαίων ε, εφόσον η Τουρκία δεν ανοίγει τα λιμάνια της για την ε, Κύπρο. Κάποια από τα κεφάλαια δεν θα προχωρήσουν επόμενο, στην επόμενη φάση των διαπραγματευσιών γιατί τα έχει μπλοκάρει η Κύπρος. Κάποια άλλα κεφάλαια δεν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση γιατί ε, τα έχει μπλοκάρει η Γαλλία. Επομένως, η δική μας δουλειά εδώ ως Επιτροπή δεν είναι να ανοίξουμε μέσα από τα μάτια των γυναικών αυτά τα κεφάλαια, γιατί είναι πραγματικά τεράστια σημασία πολιτικό θέμα και έχει και πολλές άλλες συνέπειες. Είναι θέμα πολιτικό. Προσωπικά είμαι αντίθετη για το άνοιγμα αυτού του κεφαλαίου. Ευχαριστώ. Κυρία Κώστα. Ehm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω βεβαίως ότι η κυρία Μποσκούρτ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια και η έκθεσή της είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι έχει έρθει σε άμεση επαφή με το τι γίνεται επιτόπου στην Ιταλία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια έκθεση η οποία να απεικονίζει τι συμβαίνει πραγματικά επιτόπου. Γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μποσκούρτ. Από εκεί και πέρα, ε, πρέπει να δούμε την αναλογία με τη στρατηγική για το 2020. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες προοπτικές ε, που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και την ε, γυναίκα στην Τουρκία. Γι' αυτό και εγώ παίρνω το λόγο γιατί θα ήθελα να τονίσω τα εξής σημεία. Πιστεύω καταρχάς ότι θα ήταν χρήσιμο να υπογραμμιστεί στην έκθεση η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλά κεφάλαια έχουν να κάνουν την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλά προγράμματα ε, αφορούν την Τουρκία, η κινητικότητα νέων, ε, ε, σπουδές, κατάρτιση, είσοδο στον επαγγελματικό χώρο. Επομένως θα μπορούσαμε να επιμείνουμε οι γυναίκε να διαδραματίσουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτών των εταιρικών σχέσεων. Είναι η δική μας συμβολή, ούτω ώστε να αλλάξει σιγά σιγά η νοοτροπία και να αισθανθούν οι γυναίκες ε, στην Τουρκία ε, ότι εμπλέκονται σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Εγώ ήμουν στην Κωνσταντινούπολη και παρέστην σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που είχε οργανωθεί από το Υπουργείο Αρμόδιο για τις γυναίκες και την ε, σχέση με την οικογένεια και εκεί διαπιστώσαμε με σαφήνεια ότι οι τοπικές αρχές ε, έχουν ρόλο να παίξουν και η παρουσία τους θα είναι όλο και πιο ισχυρή. Είδα δηλαδή ότι σιγά σιγά οι γυναίκες αναλαμβάνουν δεσμεύσεις στο επίπεδο της τουρκικής πολιτικής σκηνής και ενίοτε διαπιστώνουν μια κάποια έλλειψη αλληλεγγύης εναντίον τους οι γυναίκες στην Τουρκία από την πλευρά των Ευρωπαίων, της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής και κυρίως των Ευρωπαίων γυναικών. Ίσως δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο απαιτητικοί ως προς τα κριτήρια. Θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν είναι σκοπός μας ε, εμείς να υιοθετήσουμε μια δασκαλίστικη συμπεριφορά. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες. Όλοι επιθυμούμε περισσότερο εκδημοκρατισμό και σύσφυξη των σχέσεων με τις γυναίκες στην Τουρκία. Με ενδιαφέρει επίσης το θέμα της ε, απασχόλησης. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό των γυναικών ε, αυτό το οποίο δουλεύει. Επομένως δεν έχουν μεγάλη αυτονομία και λείπουν πάρα πολλές υπηρεσίες, υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Στόχος είναι να ενισχύσουμε π.χ. τις δυνατότητες μερικής απασχόλησης μέχρι ότου υπάρξουν κατάλληλες δομές για την φύλαξη των παιδιών. Και νομίζω ότι και η προηγούμενη συνάδελφος το είπε, Σίγουρα οι ανάγκε εκπαίδευση ή κατάτηση είναι πολύ μεγάλε. Η καταρτιση ειναι πολυ μεγαλε η τουρκικη αναπτύσσεται και μα εκπλήσει το γεγονό ότι διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκε δεν συμμετέχουν τόσο ενεργά όσο θα μπορούσαν στην αγορά εργασία. Βεβαίω αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση, αλλά οφείλεται και στην έλλειψη της ε, κατάρτισή τους και τη προσαρμογή τους στην αγορά εργασία. Άλλο στοιχείο εξίσου σημαντικό κατά την άποψή μου και θα ήθελα να το συμπεριλάβει η έκθεση είναι βεβαίως το θέμα ε, των εγκλημάτων, των καταναγκαστικών γάμων και των εγκλημάτων τιμής. Αυτά αναφέρονται στην έκθεση, ωστόσο να επιμένουμε περισσότερο στον ε, θρησκευτικό πλουραλισμό. Για παράδειγμα, από ό,τι φαίνεται, οι γυναίκες που δεν είναι μουσουλμάνες ε, συνεχίζουν να δυσκολεύονται ε, να συνάψουν γάμο με άτομα που έχουν διαφορετική θρησκευτική πίστη από τις ίδιες. Δηλαδή υπάρχουν επιπρόσθετες δυσκολίες ε, ως προς τη σχέση, την απρόσκοπτη σχέση μεταξύ ε, πολιτισμικών διαφορών και θρησκευτικών δογμάτων. Η κυρία Κράτσα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την κυρία Μποσκούρτ η οποία με την έκθεσή της σειρά ετών τώρα μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τη σημερινή κατάσταση και για τις προοπτικές και να συνειδητοποιήσουμε τις πολιτικές μας ευθύνε για το θέμα αυτό. Ε, πιστεύω ότι έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο αυτή η έκθεση διότι η Τουρκία ως υποψήφιο μέλος της Ένωσης συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε το ρόλο που παίζει και το θέμα των γυναικών, διότι μη γελιόμαστε, η κατάσταση των γυναικών εκφράζει το επίπεδο δημοκρατίας και πολιτισμού και, και ε, ενσωμάτωσης των, των, ε, των αρχών, των παγκόσμιων αρχών για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις χώρες που είναι προοδευμένες υπάρχει και ένα καλό επίπεδο εφαρμογής αυτών των αρχών και στις χώρες που έχουν ευρύτερα προβλήματα υπάρχει και το πρόβλημα των γυναικών. Λοιπόν, η Τουρκία πρέπει να το δει σοβαρά το θέμα αυτό γιατί συνδέεται με την πορεία της του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι όχι μόνο για τη δική της συνοχή και ευημερία αλλά και για την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η Τουρκία σήμερα φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο μοντέλου στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης και έχει μεγάλη ευθύνη στο είδος του μοντέλου που προβάλλει. Εγώ, επειδή θα έχω την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, μαζί με συναδέλφους, θα λάβω μέρος στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρατήρηση των εκλογών στην Ισία, και ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφές με την κοινωνία των πολιτών, με πολιτικούς, γυναίκες, άντρες στην Τινησία. Εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες για αν η Τουρκία μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του μοντέλου, διότι στην Τινησία που ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών πιστεύουν ότι η Τουρκία προβάλλει σε ένα μοντέλο που είναι πιστογύρισμα για αυτούς. Λοιπόν, είναι καλό αν η Τουρκία μπορεί να προβάλλει ε, ε, σήμερα να διαδώσει ένα μήνυμα στον αραβικό κόσμο εξυγχρονισμού, σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά επειδή ακριβώς να παίξει αυτό το ρόλο έχει και μεγάλη ευθύνη. Δεύτερον, πρέπει να δούμε με την έκθεση της κυρίας Μποσκούρτ με όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχει μέσα για την κατάσταση σημερινή και για αυτά που πρέπει να γίνουν, πρέπει να δούμε ότι οι ευθύνε είναι μοιρασμένε. Καταρχάς, δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, νομοθεσία και εφαρμογή της νομοθεσίας, ήδη το ότι παίρνετε μια νομοθεσία είναι ένα σοβαρό βήμα. Διότι υπάρχουν αντιστάσεις λόγω πολιτισμικών ε, μοντέλων και μέσα στην Εθνοσυνέλευση τουρκική. Το ότι καταφέρονται και ψηφίζεται ένας νόμος είναι ένα βήμα. Σοβαρό που πρέπει να το χαιρετήσουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πού είναι ευθύνε στην εφαρμογή. Παίζει το ρόλο του το εκπαιδευτικό σύστημα ε, ενημερώνονται οι δικαστές, οι αστυνομικές αρχές, ε, η ενθαρρύνεται η κοινωνία των πολιτών να κάνει καμπάνια για την ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματά τους. Είναι θέματα σοβαρά που πρέπει να τα δούμε. Θέλουμε με αυτή την έκθεση να προσφέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τον απολογισμό που πρέπει, παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων, τον ποιοτικό και τον ποσοτικό απολογισμό στη συνεργασία της με τις αρχές. Χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σοβαρή έκθεση απολογιστική και δεύτερον πρέπει να δούμε ε, επίσης πόσο το, πώς λειτουργεί το λαϊκό κράτος και πόσο η Εκκλησία αναμειγνύεται, οι θρησκευτικέ κοινότητε ή δεν αναμειγνύονται και πόσο ο ρόλος τους είναι προς την κατεύθυνση του σεβασμού των αρχών ενό λαϊκού κράτους όπου δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ε, θρησκευτική ή ιδεολογική για την ε, μη καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών και πρέπει να δούμε και ο λόγος αυτός ο θρησκευτικός ποιος είναι μέσα στην Τουρκία. Και δεύτερον είναι πολύ σημαντικό στην προσέγγιση που κάνουμε να μην παίρνουμε για να μην εστιαστούμε μόνο στα καλά παραδείγματα τις γυναίκες στην Τουρκία, επιχειρηματίες, επιστήμονες, τραπεζίτες που είναι στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα και να μην δώσουμε τη σημασία στο χάος στην κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών, κυρίως στις κουρδικές περιοχές, που επικρατεί στην υπόλοιπη Τουρκία. Μια χώρα προς ε, ένταξη υποψήφια οφείλει να υπηρετήσει μια συνοχή και μια ευημερία του συνόλου και όχι μόνο κάποια φωτεινά παραδείγματα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μποσκούρτ ε, και να είμαστε όλοι προσεκτικοί στο να εκφράσουμε ένα ελπιδοφόρο αλλά ουσιαστικό μήνυμα και απέτηση τόσο από την Τουρκία όσο και από τις ε, ευρωπαϊκές αρχές. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτή την πολύ λεπτομερή έκθεση η εισηγήτρια έχει υπογραμμίσει τα θέματα τα πιο σημαντικά και το είπαν και οι προηγούμενες ομιλήτριες. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει στην Τουρκία, δεν έχει υπάρξει βελτίωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα ανησυχητικά σήματα στην έκθεση την παγκόσμια για το 2009. όπου η, Τουρκία τοποθετείται στη θέση 129 από τις συνολικά 134. Λιγότερο από ε- το 1% των κοινοτήτων στην ε, Τουρκία έχουν ε, γυναίκα δήμαρχο. Η κυρία Μποσκούρ είναι πολύ ακριβή στην έκθεσή, τους, στην έκθεσή της. Έχει μεταβεί επιτόπου επανειλημμένος, έχει έρθει σε επαφή με τις γυναίκες στην Τουρκία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, η ιδέα θεσμοθέτησης ποσοστώσεων για τις γυναίκες θα μπορούσε να είναι μια λύση, να έχουμε ποσοστώσεις και στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι χρήσιμο βεβαίως να κάνουμε ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τις εκλογές στην Πολωνία είδαμε ότι πάρα πολλές ε, γυναίκες ήταν υποψήφιες ακριβώς χάρη σε αυτές τις ποσοστώσεις. Εγώ ανέκαθεν ε, θεωρούσα ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μπορεί να είναι και χρήσιμο εργαλείο για την περίπτωση της Τουρκίας για να μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετάσχουν περισσότερο ε, στα κοινά. Αν ισχύει αυτός ο αριθμός, δείχνει ότι οι γυναίκες είναι τελείως απούσες από την πολιτική σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονό δηλαδή ότι λιγότερο από το 1% των ε, δημάρχων σε κοινότητε είναι γυναίκε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετικά ποιοτική και δείχνει πόσο έχει δεσμευτεί η συγγήτρια να απεικονίσει την πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι εξαιρετική η έκθεση και τονίζει τα πιο σημαντικά ε, θέματα. Καταναγκαστική γάμη, για παράδειγμα. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. Όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες χώρες όπου ε, ο πληθυσμός με καταγωγή από την Τουρκία είναι αρκετά ισχυρός, αρκετά μεγάλος. Ή η βία κατά των γυναικών. Όλα αυτά τονίζονται στην έκθεση. Από την άλλη η έκθεση είναι ισορροπημένη διότι επισημαίνει ότι έχουν, έχει σημειωθεί πρόοδος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ποσοστώσεις ε, στα πανεπιστήμια σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Όμως στην Τουρκία υπάρχει ποσόστοση υπέρ των γυναικών. Ενδεχομένως λοιπόν και εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να διδαχθούμε από την τουρκική νομοθεσία. Έχουμε και την εκπαίδευση των αστυνομικών οργάνων. Εκεί η Τουρκία έχει θεσμοθετήσει κάποια μέτρα πολύ σημαντικά και οι υπόλοιπες χώρες μπορούν να εμπνευστούν από αυτά. Παρ' όλα αυτά, η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά είναι πολύ σημαντική. Θα μπορούσε να λυθεί το θέμα με την ε, θέσπιση ποσόστοσης. Και σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας και το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα συνδικάτα. Αυτό μας εκπλήττει. Αντίθετα με το τι συμβαίνει ε, στη Δανία, τη χώρα μου, στην Τουρκία πάρα πολλές γυναίκες ε, συμμετέχουν στις ε, οργανώσεις των εργοδοτών ενώ στην Τουρκία δηλαδή οι γυναίκες επιχειρηματίες οργανώνονται και εντάσσονται σε σωματεία και έτσι έχουν περισσότερες δυνατότητες να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα πρέπει να εξετάζουμε την Τουρκία, την Τουρκία ως ένα εργαλείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμπλουτίζει τη διεύρυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Κλάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Ε, πω, δεν υπάρχει πιο έγκαιρη στιγμή για να κάνουμε μια τέτοια έκθεση και είναι ιδιαίτερα σημαντική και πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούσαμε πολλές παρεμβάσει, ε, μιλούμε για μια υποψήφια χώρα προ ένταξη. Mm. Μιλούμε για διαπραγματεύσεις που τρέχουν. Και ε, το να είμαστε έτσι πολύ διπλωμάτες και λίγο ε, έτσι χωρίς να έχουμε οξύες ε, γωνίες στην, ε, στην ε, έκφρασή μας δεν νομίζω ότι μας βοηθάει. Αφόσον ε, είμαστε αυστηροί με τις άλλες χώρες πρέπει να είμαστε και αυστηροί και με μια τέτοια χώρα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερα δεδομένα και να κάνουμε πολύ περισσότερη κριτική. Ας πούμε, η, Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση λέει ότι έχει πολιτική μηδενική ανοχή της βίας κατά των γυναικών. Αυτό είναι βασική ουσιώδης απόφαση την οποία πρέπει να ε, επικρίνουμε εφόσον ακόμα υπάρχουν περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο άμεσοι, πολύ πιο συγκεκριμένοι ή λέει ότι ζητάμε από την, ε, από την Τουρκία να ποινικοποιήσει τους καταναγκαστικούς γάμους. Προφανώς, αλλά θα πρέπει και πιο πριν να πούμε κάτι. Θα πρέπει και από πριν να προετοιμάσουμε με κάποιο τρόπο το έδαφος. Δηλαδή λείπει κάτι, η εκπαίδευση, η μόρφωση, όλα αυτά πρέπει να τα, να τα τονίσουμε. Εμείς επικεντρωνόμαστε στις γυναίκες. Ξέρουμε ότι μόνο Ελάχιστε είναι οι δυνατότητες των γυναικών. Ούτω ή ο τρόπος που μεγαλώνουν οι άντρε και οι γυναίκε στην Τουρκία είναι τελείως διαφορετικές. οι πατριαρχικέ οικογένειε είναι κατά κύριο λόγο το είδο οικογενειών της Τουρκίας. Και αυτό συμβαίνει εδώ και γενιές, πολλέ γενιέ. Οπότε, ίσω σε ένα σημείο κάπου στην έκθεση θα πρέπει να πούμε ότι και τα αγόρια και τα κορίτσια θα πρέπει να πηγαίνουν σε κοινό σχολείο και να έχουν ίσα δικαιώματα, γιατί είναι ίσοι και οι άντρες με τις γυναίκες. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μπορέσουμε να ελέγξουμε ή τέλο πάντων να προτείνουμε το τι θα πρέπει να γίνεται στα σχολεία. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και για να μπορέσουμε έτσι να επιτύχουμε και κάτι μακροπρόθεσμα. Η καταναγκαστική γάμη ελάχιστε φορέ πάνε στο δικαστήριο. Προφανώς είναι δύσκολο να πάει κανένα στην οικογένειά του στο δικαστήριο και εφόσον έχει αποφασίσει τώρα πια η οικογένεια για το τι θα γίνει με, το, με, την, με την κόρη που παντρεύτηκε χωρίς ε, τη θέλησή της. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το σημείο αυτό και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Η Επιτροπή Γυναικών λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να τα πει τα πράγματα στα ράτα πρέπει να τα πούμε με το όνομά τους και γι' αυτό σας ζητώ να ε, τονίσουμε περισσότερο και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Okay. Jag vill Ευχαριστώ. Synpunkter och eh, innan jag ger ordet till eh, Mrs. Boscourt eh, för ett avslutningsord så vill jag först ge ordet till Mr. Makridis från European Commission. Κυρία Μποσκούρτ, Α, όχι, Κομισιόν πρώτα. Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό για την ένταξη της Τουρκίας και για το πώς βλέπουν την Τουρκία στην Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι γενικά Συμμεριζόμαστε την ανάλυση της κυρίας Μποσκιούρτ για τα τέσσερα κύρια θέματα όπου πρέπει να σημειωθούν πρόοδοι, δηλαδή απασχόληση, παιδεία, πολιτική εκπροσώπηση και βία κατά των γυναικών. Η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα, θετική Δεν είναι εύκολο να λύσει κανείς αυτά τα προβλήματα, χρειάζεται κάποιος χρόνος και πρέπει να δούμε και τη δυναμική των πραγμάτων. Θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή ε, λέει τα πράγματα με το όνομά τους αλλά επίσης τονίζει τομείς όπου η τουρκική κοινωνία των πολιτών, οι τουρκικές αρχές όλοι οι Τούρκοι γενικά πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να μεταφραστεί η νομοθεσία σε πραγματικότητα. Αν υπάρχει καμία συγκεκριμένη απορία να σας τη λύσω ευχαρίστως, αλλιώς δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Παπαδοπούλου. Έχω μια απορία να μου λύσει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Δεν ξέρω αν ήταν σωστή η μετάφραση. Αλλά είπατε ότι δεν είναι εύκολο να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, αναγκαστική γάμη για πολύ νεαρές κοπέλες. Κλίματα τιμής. Για όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία όχι βέβαια πολύ λεπτομερή δυστυχώ, αλλά στο Συμβούλιο της Ευρώπης άμα ψάξει κανείς διάφορες εκθέσεις του βλέπει ότι τονίζονται πολλά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσετε γιατί θεωρείτε ότι δεν είναι εύκολο να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί είναι προβλήματα που αναφέρονται επί πολλές δεκαετίες ήδη. Είναι ζωτικό λοιπόν η Κομισιόν να πάρει μια στεναρή θέση και στάση να τηρήσει. Και πέρυσι και πρόπερσι ακούστηκαν πολλά για αυτά τα θέματα και αν δεν πάρετε στεναρή θέση και στάση, τηρήσετε, θα τα συζητάμε και για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό δεν είναι σωστό. Αν θέλει η Τουρκία να μπει στην Ένωση πρέπει να σημειωθούν πρόοδοι όχι μόνο στα χαρτιά και στην νομοθεσία αλλά να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ένωσης. Εμείς δεν βλέπουμε να εφαρμόζονται αυτές οι υποχρεώσεις για τις γυναίκες. Δεν έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο ούτε έχει σεβαστεί τις υποχρεώσεις της και για τη χώρα μου την Κύπρο. Ακόμη λοιπόν και αν αλλάζει την νομοθεσία δεν σημαίνει ότι θα κάνουν πράγματι αυτά που πρέπει να κάνουν για να γίνουν μέλη της Ένωσης. Θέλω πολύ συγκεκριμένη απάντηση για αυτά. please. Μακρίδης. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ένα παράδειγμα. Υπάρχει το νομοσχέδιο για την προστασία της οικογενείας του 98 και το 7 διευρύνθηκε. Τώρα διαβάσαμε στον τύπο ότι θα ξαναδιατροποποιηθεί για να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το εύρος στο πεδίο εφαρμογής του. Θα δούμε τι ακριβώς αλλαγές θα είναι αυτές. Αλλά όταν είπα δεν είναι εύκολο να ληφθούν αυτά εννοούσα ότι το θέμα δεν είναι ακριβώς, δεν είναι μόνο να εγκρίνονται νομοσχέδια και να εφαρμόζονται διοικητικά και δικαστικά, αλλά πρέπει να γίνει και μια κοινωνική μετατροπή. Αυτή η διαδικασία δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να δούμε τη δυναμική και να ενθαρρύνουμε τη διαδικασία αυτή αλλαγή νοοτροπιών δηλαδή, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην Τουρκία που θέλουν να γίνουν αλλαγές να ενθαρρυνθούν να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία των αρχών με την κοινωνία των πολιτών ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα απτά ως το δυνατόν συντομότερα. Κάνουμε την, επιτηρούμε την κατάσταση στην Τουρκία και γνωρίζουμε γενικά με τις ετήσιες μας εκθέσεις ποια είναι η πρόοδος. Αύριο μάλιστα θα δημοσιευτεί η επόμενη ετήσια έκθεση πρόοδου για την Τουρκία. Πάντοτε προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα αντικειμενικά και για το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών και για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή ότι δεν είναι μόνο θέμα έγκρισης νομοθεσίας, ούτε μόνο διοικητικής και δικαστικής εφαρμογής, αλλά και θέμα κοινωνικής μετατροπής και αλλαγής νοοτροπίας. Αυτό το λέει η κυρία Μποσκιουρτ στην έκθεσή της. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Οπότε να δώσουμε το λόγο τώρα στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους αδελφούς για τα σχόλιά τους και για την στήριξή τους. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα θέματα που έθεσαν. Χαίρομαι για την στήριξη της πολιτικής μηδενικής ανοχής, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πολιτική κλειδί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών. Ναι. Η έκθεσή μου δεν μιλάει για το, νομοθεσία, μιλάει για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε και πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα και να γίνει κατανοητή αυτή η πολιτική. Αυτό είναι σαφές από την έκθεσή μου. Το θέμα των εγκλημάτων τιμής επίσης αναφέρθηκε από δύο συναδέλφους. Θα πρέπει όντως να γίνει πιο συγκεκριμένο στην έκθεση, οπότε θα περιμένω τις ε, προτάσεις σας για να υπάρξει μια παράγραφος σχετική. Το θέμα του προπολογισμού, το είπε και η κυρία Μάισνερ. Γι' αυτό πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών στην Τουρκία για να ζητήσω πληροφορίες, γιατί όλοι μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικές στρατηγικές και προγράμματα δράσης και νομοθεσίες και ό,τι άλλο θέλετε, αλλά χωρίς προπολογισμό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι. Επίσης, τα χρήματα που χρειάζονται, ειδικά για την αντιμετώπιση της βίας, θα είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ότι δηλαδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ισχυρή τάση κατά της βίας. Για μας είναι σημαντικό που η Τουρκία κάνει κάτι, αλλά και η τουρκική κοινωνία επίσης έχει ε, βαρεθεί να βλέπει τέτοιες περιπτώσεις, ε, τέτοια περιστατικά βίας. Και αυτό είναι σημαντικό. Το θέμα τώρα της εκπαίδευσης. Δεν μιλούμε για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το είπε και η Μπρίτα. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε πολλές ειδικότητες υπάρχουν ε, περισσότερα κορίτσια από ότι αγόρια αλλά η επαγγελματική κατάρτιση είναι επίσης πολύ σημαντική. Στην Τουρκία βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη όχι μόνο γυναικών, αλλά και αντρών για επαγγελματική, για θέσει επαγγελματική κατάρτιση. Αυτό, κατάρτισης, αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Και βεβαίω ειδικά για τι γυναίκε. Δεν το ανέφερα στην εκθεσία μου γιατί δεν μπορούσα, αλλά για τις γυναίκες α πούμε που βρίσκονται σε άσυλο έχω επισκεφθεί πάρα πολλά πάρα πολλές εγκαταστάσεις και αυτό που μου είπαν οι γυναίκες είναι ότι θέλουμε να δουλέψουμε, θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να φροντίζουμε τα παιδιά μας και θέλουν να μάθουν, να μάθουν ένα επάγγελμα ώστε να μπορούν να δουλέψουμε. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα μεν, αλλά θα πρέπει να είναι πιο ευρεία, πιο πολλά, έτσι ώστε οι γυναίκε αυτές να μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιες τον εαυτό του για να είναι ανεξάρτητες από το σύζυγό τους. Αυτό είναι σημαντικό για να βελτιωθεί η κατάσταση απέναντι στη βία. Τώρα, το θέμα των ασύλων. Ναι, στην έκθεσή μου είναι σαφές ότι θέλω να υπάρξουν περισσότερα. Ε, αν δείτε το Συμβούλιο της ε, Ευρώπης, στην ε, Τουρκία υπάρχει ο, η ίδια ε, νομοθεσία υπάρχει, ναι, πρέπει να υπάρχει μάλλον ένα άσυλο για κάθε 50.000 ανθρώπους. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει. Και το συζήτησα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και των Ιστορικών και μου είπαν ότι θα υπάρξει μια δευτερεύουσα ε, νομική πράξη που θα ε, εφαρμόζει αυτό το νόμο, ότι δηλαδή θα υπάρξουν περισσότερα άσυλα. Ας πούμε, ε, στην ε, Τουρκία τώρα θα έπρεπε να υπάρχουν 200 παραπάνω άσυλα και δεν ισχύει, δεν υπάρχουν. Τώρα, το θέμα του κεφαλαίου 23. Νομίζω ότι όντω είναι ουσιώδου σημασία γιατί μιλούμε για θεμελιώδει αξίε. Αν θέλουμε ω Ευρώπη να έχουμε δυνατότητα μόχλευση, πίεση στην ε, Τουρκία, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μιλήσει ακριβώ για αυτά, για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι αξίε δεν έχει μπλοκαριστεί λόγω του επιπλέον, ε, του επιπλέον πρωτοκόλου. Έχει μπλοκαριστεί λόγω διμερών ε, θεμάτων που προκύπτουν με την Κύπρο το κεφάλαιο αυτό. Οπότε για το κεφάλαιο αυτό, για το θέμα μάλλον αυτό, οι γυναίκες της ε, Τουρκίας όντως ε, πρέπει να τύχουν καλύτερων θεμελιωδών δικαιωμάτων, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και το τονίζω και στην έκθεσή μου. Για το θέμα των γυναικών στην πολιτική, το είπε και η συνάδελφος, ναι. Σημαντικό σημείο. Στις τελευταίες ε, εκλογές είχαμε 14% συμμετοχή γυναικών. Προφανώς πρέπει το ποσοστό αυτό να αυξηθεί. Αλλά νομίζω ότι και μεταξύ Ευρώπης και ε, η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας στο θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντική. Η κυρία Κράτσα επίση είπε κάτι σημαντικό, ότι η Τουρκία μπορεί να είναι μοντέλο για τα, για τα δικαιώματα των γυναικών σε ό,τι αφορά τι αραβικέ χώρε. Το στηρίζω αυτό, συμφωνώ όντω μπορεί να βοηθήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στι χώρε αυτέ. Η Μπρέτα Τόμσον είπε ότι μίλησε για το θέμα των ε, αναγκαστικών γάμων. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, οι αναγκαστικοί γάμοι απαγορεύονται στην Τουρκία αλλά δεν βρίσκονται ως, δεν ποινικοποιούνται από το ποινικό δίκαιο. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι να μπουν στο ποινικό δίκαιο και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Άκουσα και μια ιστορία από μη κυβερνητικέ οργανώσει που λέει ότι ένα κορίτσι υποχρεώθηκε να παντρευτεί έναν άντρα, υποχρεώθηκε από την οικογένειά της, δεν ήθελε να τον παντρευτεί και έμαθε ότι υπήρχαν κάποια μαθήματα στο, σε μια τοπική σχολή και τη είπαν ότι μπορούσε. Α, συγγνώμη, ότι ε, υπήρχε ένα δικαστήριο το οποίο μπορούσε, στο οποίο μπορούσε να πάει και να πει ότι με υποχρέωσαν να παντρευτώ. Και πήγε στην οικογένειά της ίδια και είπε ότι εγώ, ε, μπορεί, να με υποχρεώνετε, αλλά εγώ θα πάω στο δικαστήριο για να ακυρώσω το γάμο αυτό και τελικά αυτό αρκούσε αυτή η απειλή για να κάνει πίσω η οικογένεια και να μην την υποχρεώσει να παντρευτεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι γυναίκε ε, για τα δικαιώματά τους. Είναι σημαντικό, ε, ειδικά για τις χώρες της Ανατολικής Τουρκίας που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πολλές γυναίκες έχουν δικαιώματα, αλλά δεν τα ξέρουν. Τα συνδικάτα τώρα. Ε, Όντω είναι ανησυχητικό παράγοντα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Τουρκία να γίνει κάποιο μέλο ε, συνδικάτου, είτε είναι άντρα είτε είναι γυναίκα. Αν είναι και γυναίκα, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Υπάρχουν ε, επιπλέον προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει ε, μέλος. Τώρα για το θέμα της εκπαίδευσης και για τα αγόρια, ναι, σημαντικό, το λέω και εγώ στην ε, έκθεσή μου ότι θα πρέπει και τα αγόρια και τα κορίτσια να συμπεριλαμβάνονται. σε αυτούς που μπορούν να ε, τύχουν ε, εκπαίδευσης. Γι' αυτό μιλάω για ισότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και την εκπαίδευση των αγοριών πέραν του θέματος της εκπαίδευση των κοριτσιών. Βεβαίως, χαίρομαι πολύ για τα σχόλιά σας και προσβλέπω στις, στη συμβολή σας και στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Okay, um, okay, please. Very, very short correction. There are... Μία σύντομη διορθωσούλα. Opening of chapter 23 is not a bilateral issue. Δεν είναι διμερές θέμα η συμφωνία που αναφέρθηκε. Δεν έχουν διμερείς σχέσεις η Κύπρος και η Τουρκία γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη δημοκρατία της Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία διμερή σχέση λοιπόν. Το θέμα είναι μόνο μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας, όχι Κύπρου και Τουρκίας. Αυτό να το αποσαφηνίσουμε γιατί έτσι είναι τα πράγματα και έχω εδώ και το σχετικό έγγραφο. Δεν είναι θέμα Τουρκίας και Κύπρου. Ορίστε. Okej, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μποσκούρτ για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ και όλες όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση και όλους επίσης. Τώρα, κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η Επιτροπή θα ψηφίσει στις 21 και 22 Νοεμβρίου και θα εξεταστεί το θέμα στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου του 2012. Αυτά για το θέμα αυτό. Περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Στρέλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ θα ασχοληθούμε με μία έκθεση η οποία απευθύνεται στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων. Αυτή η Επιτροπή, Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα επί της ουσίας. Είναι σύντομο το έγγραφο αυτό, περιλαμβάνει μόνο πέντε σημεία, έχουμε όμως συμπεριλάβει τα ουσιώδη, πιστεύω. Όπως γνωρίζετε, οι γυναίκες προτιμούν να επιλέγουν τη μορφή του συνεταιρισμού, ε, προκειμένου να διασφαλίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά τους συμφέροντα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους επιδιώξεις ή προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται. Επίσης επιλέγουν τη συνεταιριστική μορφή για να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι συνεταιρισμοί είναι ε, μια επιχειρηματική μορφή που διέπεται κυρίως από τις αρχές της αυτοβοήθειας, ε, της αλληλεγγύης, της ευθύνης, της ισότητας μεταξύ των μελών. Τα μέλη των συνεταιρισμών βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και είναι τα μέλη αυτά καθεαυτά που προσδιορίζουν με δημοκρατικό τρόπο τις στρατηγικές ε, που θα ακολουθήσει ο συνεταιρισμός για να επιτύχουν τους στόχους τους, τους οικονομικούς, κοινωνικούς ή πολιτισμικούς. Γι' αυτό το λόγο ο συνεταιρισμός είναι ιδανική νομική μορφή, πιστεύω, για να καλυφθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες των γυναικών. Μπορεί κανείς να έχει ε, αποκλειστικά γυναικείους συνεταιρισμούς, αμυγός γυναικείους ή και μικτούς. Η συνεταιριστική, συνεταιριστική μορφή δίνει στις γυναίκες μέλη ή εργαζόμενες στους συνεταιρισμούς, τους δίνει δυνατότητες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, διότι θα έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία, σε ε, ιδρύματα αποταμίευσης, σε υπηρεσίες ε, κατοικίας, ε, εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες κατάρτισης. Είναι θετικά όλα αυτά. Έχουμε όμως και ένα ε, αρνητικό, διότι πάντοτε το νόμισμα έχει δύο πλευρές. Οι συνεταιρισμοί δεν διαφοροποιούνται από τις άλλες εταιρικές μορφές. Δηλαδή και σε ένα συνεταιρισμό μπορεί να έχουμε ανισότητες, οι οποίες να παραμένουν μπορεί να υπάρχουν συνεταιρισμοί που κάνουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών ως προς την πρόσβασή τους σε διευθυντικές θέσεις. Ε, και στους συνεταιρισμούς τις διευθυντικές θέσεις τις κατέχουν ε, άνδρες κατεξοχήν. Ε, αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία είναι μια δυνατότητα να έχουμε περισσότερη ισότητα στην ε, πρόσβαση στις θέσεις όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στις διαδικασίες που θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγούν όσοι θα καταλάβουν τα, ε, τις διευθυντικές ε, θέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στατιστικά στοιχεία συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών. Όμως οι γυναίκες είναι η πλειονότητα των απασχολούμενων στον κλάδο αυτό. Όπως όμως συμβαίνει και σε άλλους τομείς ε, της ε, δραστηριότητας, δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ε, στα κλιμάκια όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εκπονήσει μία μελέτη με συγκρίσιμα στοιχεία κατανεμημένα μεταξύ των δύο φύλων, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς το, τους δείκτες συμμετοχής των γυναικών στους συνεταιρισμούς. Και αυτό είναι μία από τις προτάσεις που θα βρείτε στην έκθεσή μου. Σε ορισμένους κλάδους και σε ορισμένα κράτη-μέλη ο συνεταιρισμός είναι ο βασικός παράγων για την παραγωγή, τη διανομή και την παροχή των υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Είναι εξαιρετικά σημαντικός ο συνεταιρισμός και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένες χώρες-μέλη. Ε, προωθεί τη βελτίωση των ικανοτήτων, προωθεί την εκπαίδευση ε, στις μικρές περιφερειακές κοινότητες. Η έννοια λοιπόν της ε, κατάρτισης, ε, της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης των γυναικών είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι συνεταιρισμοί βασίζονται σε αρχές και σε αξίες και γι' αυτό συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί, αυτό ε, αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Γι' αυτό και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των συνεταιρισμών και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτούς. Η εφαρμογή της οδηγίας 72 του 2003 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη, η διαδικασία εφαρμογής τη διάσταση του φύλου. Ορισμένα κράτη-μέλη συνεχίζουν να μην ε, συμμορφούνται με την οδηγία αυτή, ειδικότερα όσον αφορά την εξισορροπημένη ε, συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές που κάνουν τις διαπραγματεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασιστεί ο διορισμός των ε, υπευθύνων στις διευθυντικές θέσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη διάσταση του φύλου όταν ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά η Οδηγία 72 του 2003. Και θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη διάσταση του φύλου και ε, στην ε, ε, μελλοντική αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Έχετε το λόγο, ήδη τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Εστρέλα για την έκθεση αυτή. Είναι πολύ καλογραμμένη, δεν έχω τίποτα να προσθέσω, πράγμα πολύ σημαντικό. Ε, θέλω όμως να τονίσω δύο σημεία. Η έλλειψη ισορροπίας στις ηγετικέ θέσεις ε, στους συνεταιρισμούς είναι μια πραγματικότητα. Ακόμα και αν θεωρείτε ότι ο καλύτερος άνθρωπος για μια θέση είναι μια γυναίκα, ε, μερικές φορές αυτό αποφεύγεται. Και είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη, σε αρκετά καλή μέλη. Ακόμα και στα κράτη-μέλη που παραδοσιακά έχουν προωθήσει ε, την ισότητα των δύο φύλων. Δεύτερη παρατηρήση οι γυναίκες να είναι πιο παρούσες στο επιχειρήν. Αυτό είναι καλό, βέβαια. Ωστόσο, θα πρέπει η Επιτροπή να εξετάζει προσεκτικά, αλλά και οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς να εξετάζουν προσεκτικά πόσο δυσκολεύονται να διεκδικήσουν ε, τις ε, ε, θέσεις ευθύνης. Δεν έχω καμία τροπολογία να υποβάλω, εκφράζω την πλήρη στήριξή μου στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί μας παρουσίασε κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ουσιώδη. Ε, οφείλω να υπεθυμίσω δύο στοιχεία. Πρόσφατα συμμετείχα σε μια συνεδρίαση συντονιστριών ε, γυναικών ε, που είχε να κάνει με τον κόσμο των συνεταιρισμών των συνεταιρισμών στην Ιταλία. Ε, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Η Επιτροπή μας μπορεί να βοηθήσει ώστε να ενισχυθεί και να στηριχθεί ε, η γυναίκα που λειτουργεί συντονιστικά σε επίπεδο ομοσπονδίας συνεταιρισμών σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή οι συντονίστριες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, είναι παρούσες Πολύ συχνά σε εθνικές ομοσπονδίες η συντονίστρια ε, των κατατόπους συνεταιρισμών είναι γυναίκα. Και είναι χρήσιμο λοιπόν να αναδείξουμε τον ρόλο ε, των γυναικών που λειτουργούν συντονιστικά μεταξύ των διαφόρων συνεταιρισμών. Δεύτερον, έχει γίνει μια ανάλυση για τα θέματα αυτά στην Αταλία και έχει δείξει, έχει καταδείξει ότι οι γυναίκες παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο και οι συνεταιρισμοί είναι ε, οι ενότητες που έχουν πληγεί λιγότερο από την παρούσα κρίση και δύναται να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Να αναδείξουμε λοιπόν αυτή την ανάλυση, να δείξουμε ότι ο κόσμος της συνεργασίας είναι αυτό που αντιστέκεται περισσότερο στην ανεργία των γυναικών και μπορεί να δώσει επαγγελματικές διεξόδους τουλάχιστον για το ξεκίνημα. Από εκεί και πέρα κάτι πιο συγκεκριμένο τώρα, κατά την άποψή μου, οφείλουμε να διαπιστώσουμε το εξής. Οι γυναίκες συμμετέχουν στους συνεταιρισμούς, αλλά δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στις ομάδες που έχουν επιφορτιστεί με τη διαπραγμάτευση. Ποια κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία δεν συμμορφούνται με την Οδηγία 72. Το ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούν τα ονόματα των χωρών για να είμαστε όλοι καλύτερα ενημερωμένοι. Συν της άλλης, θα ήταν καλό να ζητήσουμε το εξής να δοθεί περισσότερη προσοχή στην παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού ε, του 2009 για την ε, κοινωνική οικονομία. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν μέρος της κοινωνικής οικονομίας. Και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη και την ε, Επιτροπή να εντάξουν την κοινωνική οικονομία σε όλες τις ε, πολιτικές που βοηθούν στην ενίσχυση της απασχόλησης. Ο κανονισμός λοιπόν δεν έχει ε, εφαρμοστεί στην πράξη, είναι νεκρό γράμμα ουσιαστικά και θα πρέπει να ζητήσουμε ε, την ε, εφαρμογή του. Κυρία Κράτσα. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα κι εγώ με όλο το πνεύμα το οποίο έχει εκφραστεί και από τη γνωμοδότηση της κυρίας Εστρέλα και από τις ε, παρατηρήσεις και συμπληρώσεις των συναδέλφων. Είναι πολύ σημαντικό να μην πέσουμε στην παγίδα που λέει ότι οι γυναίκες είναι παρούσες στους συνεταιρισμούς. Πράγματι υπάρχουν γυναίκες. Υπάρχουν και συνεταιρισμοί γυναικοί εμείς θέλουμε και αυτό το μοντέλο να ενθαρρυνθεί, είναι άλλη κατηγορίας πρόβλημα, το συνεταιρίζεσθε των γυναικών, αλλά από την άλλη πλευρά να έχουν μια ανταγωνιστική παρουσία σε όλα τα επίπεδα οι γυναίκες, σε όλο το, θέμα, σε όλο το φάσμα των συνεταιρισμών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε στοιχεία απολογισμό ποιοτικό και ποσοτικό, να δούμε δηλαδή εκεί που ποια τα κράτη-μέλη που έχουν τα δυσκολότερα προβλήματα εφαρμογής της ε, οδηγία και του κανονισμού των σχετικών ποια, α, και πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα. Ε, είναι εύκολο να λέμε ότι δεν είναι δραστηριοποιημένες οι γυναίκες αλλά πρέπει να δούμε και το ρόλο που παίζουν οι ε, εθνικές ε, αρμόδιες αρχές. Εάν οι ίδιες έχουν τη μέρη να ενημερωθούν οι γυναίκες, να ενημερωθούν όλοι οι υπεύθυνοι του κινήματος για το ρόλο που πρέπει να έχουν οι, οι, γυναίκες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους στόχους που πρέπει να υπηρετήσει το συνεταιριστικό κίνημα. Γι' αυτό ελάχιστα πράγματα έχω να συμπληρώσω, κάποιες διευκρινήσεις ε, εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας βάσει ε, σε, αυτή την κατεύθυνση της ε, διευκρίνησης και της ανάγκης πια να έχουμε ένα σοβαρό ποιοτικό και ποσοτικό ε, απολογισμό και ε, μια μέθοδο εργασίας. Αποδεικνύεται ότι τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για το θέμα αυτό που εμπεριέχονται και οι εθνικές αρχές παίζουν ρόλο ε, πρέπει να έχουμε ένα, ένα action plan, μια μέθοδο που θα βοηθήσει και τους ίδιους τους συνεταιρισμούς και τις ίδιες τις αρχές να εφαρμόσουν την οδηγία και τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Tack för Och då innan jag ger ordet... καλά. Κυρία Εστρέλα, θα σας δώσω το λόγο, αλλά προηγουμένως θέλω να δω αν η Κομισιόν έχει να προσθέσει τίποτα. Δεν ξέρω ποιος την εκπροσωπεί εδώ μέσα. Ορίστε εσείς εκεί πίσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλουμε την έκθεση αυτή να τη βάλουμε, να τη θέσουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δηλαδή η οδηγία συμπληρώνει το θέμα του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού. Και τώρα γράφουμε έκθεση για το καταστατικό αυτό και θα δούμε ταυτόχρονα έτσι αν η οδηγία χρειάζεται τροποποίηση. Δεύτερον, Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Εταιρείας τον Ιούλιο κάναμε διαβουλεύσεις με τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους για να δούμε αν χρειάζεται καμία αναθεώρηση γιατί αυτά τα δύο νομοθετήματα ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία σχετίζονται έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα προβλήματα του ενός θα έχουν επιπτώσεις και επί του άλλου. Και τρίτον θέλουμε να τονίσουμε ότι προς το παρόν, το βλέπετε και στην έκθεσή μας, δεν έχουμε ακόμη αρκετή εμπειρία με ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς γιατί δεν είναι και πολλοί. Στην έκθεση αναφέρονται τα με 32 λέει εργαζομένους. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε βέβαια. Θα τα δούμε προσεκτικά και τις συστάσεις της Επιτροπής σας. Στη δική μας έκθεση αναφέρουμε ποια είναι τα κράτη-μέλη που ακόμη δεν έχουν εφαρμόσει όπως πρέπει τις ρήτρες ισότητος των φύλων και είναι η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ρουμανία και η Εσλοβακία. Αλλά όπως είπα και πριν αυτό αναφέρεται μόνο στους συνεταιρισ... στις συνεταιριστικές εταιρείε και όχι στους συνεταιρισμούς. Θα δούμε τι θα προκύψει από την ανάλυση μας. Ευχαριστώ. Tack för det. Och eh, det var, jag att ni kanske Δεν ξέρω, θέλετε και οι δύο να πείτε κάτι, όχι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στην κυρία Στρέλα. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο από τις διάφορες ομάδες και άκουσα τα σχόλιά τους. Τους ευχαριστώ όλους. Θα έχω καταγράψει ό,τι είπατε. Ε, μάλλον τα σχόλιά σας θα μεταφραστούν και σε τροπολογίες για την έκθεση. Έχω και εγώ βεβαίως κάποια σχόλια για να τροποποιήσω με κάποια, σε κάποια σημεία την έκθεσή μου. ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις πληροφορίες της και σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες για τα όσα συζητούμε σχετικά με τούτη την έκθεση. Και επίσης απαντήσατε στην ερώτηση της κυρίας Κώστα για το γιατί κάποια κρατημέλη δεν έχουν εγκρίνει και εφαρμόσει την οδηγία. Μόνο πέντε κρατημέλη τα έκαναν. Η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Μάλτα. Να απαντήσω σύντομα σε κάποια σχόλια. αν υπάρξει μια πρωτοβουλία Κοινοβουλίου του Κομισιόν για την εισαγωγή ενός συστήματος ποσοστώσεων για να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση και των δύο φύλων στην διοίκηση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών αλλά και άλλων εταιριών θα πρέπει να εφαρμόζονται και τα ίδια στάνταρ, τα ίδια μέτρα και στις μάκες στις, στους όπως είπα, οι γυναίκες ακόμη ε, έχουν να αντιμετωπίσουν ε, ανώτατα όρια εκπροσώπησης σε, και στις ενδραστικές εταιρείε και σε άλλες. Δεν τους επιτρέπεται να λάβουν ας πούμε θέσεις ευθύνη ε, ώστε να μπορούν να πάρουν αποφάσεις στους συνεταιρισμούς. Αυτό λοιπόν που θέλουμε εμείς εδώ να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σωστή εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Είτε μιλούμε για την πολιτική, είτε μιλούμε για επιχειρηματικές δραστηριότητε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τους συνεταιρισμούς, για τα cooperatives. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα όσα είπε η κυρία Κώστα, είπε ότι οι συνεταιρισμοί δεν ε, έχουν ε, νιώσει τις επιπτώσεις της κρίσης. Ε, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Μακάρι να συνέβαινε. Ίσως στην Ιταλία να συμβαίνει και αν συμβαίνει τότε καλά είναι τα νέα. Αξίζει μάλλον να το σημειώσουμε και να δούμε πώς τα κατάφεραν οι Ιταλοί. Αλλά θέλω να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε πιο πριν για τις αρχές και τις αξίες είναι πολύ σημαντικέ και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στους συνεταιρισμούς, Βεβαίω και στην κοινωνία, ειδικά όταν μιλούμε για την αντιμετώπιση τη κρίση. Η κρίση χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, ε, επιβραδύνει τις οικονομικές δραστηριότητε σε κάποια κράτη-μέλη πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτές οι αρχές και οι αξίες των συνεταιρισμών θα είναι αυτές πάνω στις οποίες θα πρέπει να βασιστούμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις προτάσεις σας, για τα σχόλιά σας. Έχω σημειώσει ό,τι είπατε και πραγματικά προσβλέπω στην έγκριση ε, μιας βελτιωμένης εκδοχής αυτής εδώ της έκθεσης ώστε να μπορέσουμε να τη στέλνουμε και στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ. Mm, Ευχαριστώ κύριε Εστρέλα για την ε, απάντησή σας. Να ευχαριστήσω και όλους όσους πήραν μέρο στη συζήτηση. Έχουμε και χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τροπολογίες 18 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι και η Επιτροπή μας θα ψηφίσει 21-22 Νοεμβρίου και μετά η ε, ψηφοφορία στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου. Οπότε, κλείνουμε το σημείο αυτό και πάμε στο σημείο 9. Η κατάσταση των ε, γυναικών σε περίοδο πολέμου. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Νικολάη, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η τελευταία μας σημερινή έκθεση, αλλά όχι και η λιγότερο σημαντική. Καταρχήν ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. 111. Πράγμα που δείχνει ότι η έκθεση δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των συναδέλφων όλες συνεισφέρουν, προσφέρουν κάτι στην έκθεση. Οι περισσότερες, στις περισσότερες ε, έδωσα σημασία χωριστά αλλά κυριέτερα στα αυτές που μιλούσαν για την σεξουαλική βία ως πολεμική τακτική την εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων τέτοιου είδους και στην παράγραφο 3 κατετέθηκαν πολλές τροπολογίες που αφορά την προώθηση του ρόλου των γυναικών στις πολεμικές δραστηριότητες και στην κυρώσεις κατά της επιβολής σεξουαλικής βίας σε γυναίκες ως ε, πολεμικής τακτικής. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε σωστά για να υπάρξουν συμβιβαστικές τροπολογίες και ότι μπορεί πράγματι να βελτιωθεί η έκθεση αυτή αν πετύχουμε αυτούς τους συμβιβασμούς. Θα ήθελα να τονίσω και μερικά πράγματα αν και δεν είναι αμφιλεγόμενα δηλαδή ότι οι μαζικοί βιασμοί ήδη αναγνωρίζονται από τη συνθήκη της Γενέβης ως έγκλημα και στο ψήφισμα 18-20 του ΟΗΕ. Το κύριο πρόβλημα εδώ είναι ότι υπάρχει ατιμορρησία. Μόνο δύο καταδίκες έχουν σημειωθεί. Μία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιγκοσλαβία και μία για την υπόθεση της Ρουάντας το 90. Δυστυχώς στις σημερινές σειράξεις σημειώνονται πολλές περιπτώσεις που δεν αναφέρονται και δεν τιμωρούνται. Αυτό είναι το πρόβλημα, η ατιμορρησία και γι' αυτόν τον λόγο ζητώ με σθένος να επιτρέπεται να παίζουν ένα ρόλο οι γυναίκες και στις ειρηνευτικές διαδικασίες ώστε να δίνεται η δυνατότητα στη δικαιοσύνη να παίξει το ρόλο της διότι δυστυχώς Ακόμη και οι δικαστές καθυστερούν και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα της ατιμορρησίας. Αυτό. Ιδιαίτερα για τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών κατά... σε περίοδο πολέμου. Ζήτησα να οργανωθεί μια συνάντηση με όλους τους κοιόδης για να κάνουμε τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες γιατί πολλές από αυτές μπορώ να τις χρησιμοποιήσω. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος, έχει, ποιος θέλει το λόγο. Η κυρία Γκαρθία Πέρες πρώτον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω επί της τελευταίας δήλωσης που έκανε η κυρία Νικολάη. Όντως ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει τη σημασία που δίνουμε σε αυτό το θέμα και δεν αποτελεί καμία αμφισβήτηση της έκθεσης ίσα ίσα. Αναφέρεται σε όλα τα σημαντικά θέματα και προβλήματα. Πρέπει όμως βέβαια να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες για να γίνει το κείμενο εύληπτο, να μην έχει αντιφάσεις και να είναι ικανοποιητικό για όλους και όλες. Είμαι στη διάθεση της εισηγητρίας για να συνεργαστώ για συμβιβασμούς. Σημερίζομαι όλες σχεδόν τις απόψεις που εκφράζει Ορισμένες τροπολογίες ζητούν τη διαγραφή ορισμένων παραγράφων. Αυτό δεν είμαι βέβαιη ότι θα βελτιώσει τα πράγματα. Νομίζω ότι πιο χρήσιμο θα ήταν να μιλάμε για τις υγειονομικές υπηρεσίες και όχι να διαγράψουμε αυτές τις παραγράφους. Εξάλλου οι γυναίκες είναι από τα πιο ευάλωτα άτομα σε περίοδο πολέμου και αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες και άρα ό,τι η υπηρεσία μπορεί να τις βοηθήσει δεν είναι περιττή. Επομένως, με αυτό το πνεύμα όλες οι τροπολογίες που μιλούν για αυτό το θέμα δεν πρέπει να καταργηθούν. Και ο ρόλος των γυναικών σε περίοδο ειρήνης είναι σημαντικός, όχι μόνο σε περίοδο παλέμου γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που είναι μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και που παίζουν σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Να επιμείνουμε επίσης να ενσωματωθούν οι γυναίκες στις διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων. Πολλές φορές έχουμε ακούσει αυτή την πρόταση, ότι αν ήταν τα χέρια γυναικών η επίλυση των συγκρούσεων, τότε Πολλοί από τους πολέμους που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη γη μας δεν θα υπήρχαν ή θα είχαν λήξει πολύ νωρίτερα. Σημαντικό λοιπόν είναι να δώσουμε κίνητρα και να στηρίξουμε τη συμμετοχή των γυναικών στις ε, διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων. Και τέλος, θα ήθελα επίσης να πω το εξής. Ε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα νέο πολύ σημαντικό και πολύ θετικό για τη δική μας Επιτροπή και για όλες τις γυναίκες γενικότερα. Όπως ξέρετε το Νόμπελ Ειρήνης το κέρδισαν τρεις γυναίκες οι οποίες ε, έχουν κάνει πολύ σημαντική δουλειά σε αυτό το τομέα. Ίσως με μια προφορική τροπολογία ή με κάποιον άλλο τρόπο να συμπεριλάβουμε μια παράγραφο η οποία θα αναφέρεται σε αυτό το, το νέο Ας ελπίσουμε να έρθει η μέρα όπου δεν θα είναι πια νέο το γεγονός ότι το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε σε τρεις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία μου κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω ε, τα συγχαρητήρια μου στην κυρία Νικολάη γιατί έχει ε, κάνει ένα πάρα πολύ καλό report. Προσωπικά έχω βάλει 14 τροπολογίες δίνοντας έφαση ακριβώς στο ψυχολο... στη ψυχολογική στήριξη που χρειάζονται οι γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική βία και οπωσδήποτε το γεγονό ότι η έκθεση αυτή καταδικάζει στεναρά τη συνεχιζόμενη χρήση σεξουαλικής βία κατά γυναικών ως τακτικής πολέμου νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η έφαση που δίνει η συγγήτρια όσον αφορά την ατιμορρησία είναι επίση σημαντική και στέκομαι σε αυτό γιατί δυστυχώ πολλέ φορέ είδαμε σε περιπτώσει πολέμου πολλές γυναίκες το έχουμε ζήσει και στη δική μου πατρίδα να έχουν ε, γίνει θύματα βιασμού σεξουαλικής παρενόχλησης ε, και δυστυχώς υπάρχει ατιμορρησία για πολλά χρόνια. Όταν η δικαιοσύνη δεν απονεμηθεί την ώρα που πρέπει και άμεσα τότε η ειρήνη δεν μπορεί να εδραιωθεί. Επομένω, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι οι δράστε πρέπει να προσάγονται στη δικαιοσύνη, να υφίστανται τι ποινικέ συνέπειε των πράξεων του και η ατιμορρησία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Και υποστηρίζω ακριβώ τη σύσταση που έχει κάνει η συγγήτρια ότι η άτυπη ομάδα εργασίας γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια πρέπει να καθιερωθεί θεσμικά και να αποκτήσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και αίτημα της Επιτροπής μας και εύχομαι αυτή η εισήγηση να περάσει. Ευχαριστώ. Eh, και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή. Ωστόσο, έχω κάποιες υποδείξεις να κάνω για τρία θέματα. Πρώτον, το εμπόριο ανθρωπίνων όντων να είναι, είναι ένα από τα εγκλήματα του πολέμου και της μεταπολεμικής περίοδου πέρα από τη σεξουαλική βία και τους βιασμούς, έχουμε και αυτή την δυστυχή πραγματικότητα, ε, η οποία πλήττει κυρίως τις γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά. Θα πρέπει να αλλάξουμε και τη διατύπωση σε μια πρόταση που υπάρχει στην έκθεση αυτή. Μιλούμε για τις ηρωίδες του πολέμου. Αλλά δεν θα πρέπει να πούμε τις ηρωίδες του πολέμου, τις ηρωίδες της διατήρησης της ειρήνης, για να μην δώσουμε λαβή για αμφιλεγόμενα σχόλια και παρατηρήσεις. Και να αναγνωρίσουμε και το έργο των γυναικών στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, το έργο που έχει να κάνει με τη διατήρηση της ειρήνης η δέσμευση, η στρατιωτική αλλά και η πολιτική θα πρέπει να είναι ίδια, να δίνουμε ίδια σημασία και στα δύο σκέλη. Πολύ συχνά οι γυναίκες λειτουργούν ως πολιτιστικές ε, μεσολαβήτριες, αν θέλετε, πολιτισμικές. Και τέλος, σας καλώ κύριε Πρόεδρε να το εξετάσετε, το θέμα αυτό, ίσως έχει ληφθεί απόφαση σε επίπεδο συντονιστών. Πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να υπογραμμίσει σαφέστατα το γεγονός ότι βεβαίως χαιρόμαστε για το βραβείο Νόμπελ που απονεμήθηκε στις ε, τρεις γυναίκες αυτές. Εγώ συμμετείχα, αυτό, συμμετείχα πολύ σε αυτή την διεθνή εκστρατεία Help Now η οποία τελικά στέφθηκε με επιτυχία. Ωστόσο, όταν η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγε στη Νέα Υόρκη, εκεί είχα ζητήσει ε, ρητά από την κυρία Ρέντιν να εκφράσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη μεγάλη εκστρατεία και η κυρία Ρέντιν δεν έδωσε καμία απάντηση. Πολλοί πήραν το λόγο ατομικά, οι μέλη ενώσεων, οι ομάδες κοινοβουλευτικές, ωστόσο δεν επιμείναμε ότι είναι μια νίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό και θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο από αυτό. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάη γιατί έκανε μια πολύ ολοκληρωμένη δουλειά Απριόρι η ομάδα του ΕΛΚ δεν θα έχει πρόβλημα με την πλειονότητα των τροπολογιών, ωστόσο προκειμένου να είναι πιο εύληπτη διατύπωση του κειμένου, καλό είναι να φτάσουμε σε όσο δυνατόν περισσότερες συμβιβαστικές λύσεις για να εγκρίνουμε όσο δυνατόν περισσότερες τροπολογίες. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να εκφραστούμε τούν οι εξής ιδέες στις συμβαστικές προτάσεις. Η καταπολέμηση της ατιμορρησίας, ε, τροπολογία 75 της κυρίας Παπαδοπούλου, να γίνει μεγάλο, μεγάλος θόρυβος αν θέλετε ως προς τις δικαστικές διώξεις για να φανεί ότι δεν είναι ανεκτές τέτοιου είδους δράσεις. Δεύτερον, ψυχολογικές και άλλες επιπτώσεις στα θύματα και στις οικογένειές τους. Τροπολογία 7, νομίζω ότι θα εγκριθεί μέσω κάποιας συμβαστικής λύσης. Τρίτον, ε, ε, περιπτώσεις ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης από πλευράς μελών της διεθνής, διεθνούς κοινότητας. Τροπολογίες 58 και 110. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αποζημίωση θυμάτων. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν στις συμβαστικές τροπολογίες. Στη συνέχεια, είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός, μιας ειδικής θέσης για τις γυναίκες την ειρήνη και τη σταθερότητα. Είμαι εναντίον της τροπολογίας 95. Και τέλος, έκτον, σε μια συμβαστική τροπολογία να συμπεριληφθούν οι τροπολογίες ε, Ζαμπόλξα και Χιμένεθ για τις γυναίκες καμικάζι και τις γυναίκες που συμμετέχουν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, δράσεις. Δεν πρόκειται για θύματα πολέμου, αλλά για θύτες πολέμου, αν θέλετε, ε, δρόντα στοιχεία τροπολογίες 28, 31 και 73. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά της. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Συμφωνώ πλήρως με τις προτάσεις σας. Και βεβαίως θέλω να συζητήσουμε τη ψυχολογική βοήθεια, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Βεβαίως να συζητήσουμε για τις γυναίκες καμικάζι, είναι μια άλλη πλευρά του νομίσματος, μια άλλη πτυχή του πολέμου. Κάποιες προτάσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες και θα τις ενσωματώσω καθεαυτές γιατί σε ορισμένες τροπολογίες είμαι έτοιμη να τις δεχθώ όπως είναι. Αλλά άλλες επειδή υπάρχουν επικαλύψεις καλό θα είναι να συνεργαστούμε για να έχουμε σωστή ε, συμβαστική λύση. Βεβαίως το τράφικιν γυναικών και παιδιών είναι πρόβλημα. Όχι όμως μόνο στις περιοχές όπου έχουμε ένοπλες συγκρούσεις. Είναι γενικότερο πρόβλημα ακόμα και αν σε μια περιοχή δεν υπάρχει πολεμική σύραξη και εγώ αυτό θέλω να το τονίσω. Τώρα, ε, το θέμα του βραβείου Νόμπελ. Γνωρίζω ε, την κυρία Τζόνσον, την ε, πρόεδρο της Λιβερίας. Είναι παράδειγμα της μάχης των γυναικών για την ειρήνη. Η, στην, η πρόεδρος της Νιγηρίας αντιμετώπισε 20 χρόνια φιλίου πολέμου η δράση της είναι γνωστή, όπως και των υπολείπων. Είναι καλό λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και για να ενθαρρύνουμε ε, τις γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα εντό εισαγωγικών. Θα τα πούμε την ε, επόμενη εβδομάδα, σας ευχαριστώ και πάλι, για να δούμε ποιες ε, θα είναι οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Και εμεί σας ευχαριστούμε κυρία Νικολάου που αναλάβατε αυτή την έκθεση και εσείς και όλοι οι άλλοι τη φροντίζετε με μεγάλη ορμή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι θα ψηφίσουμε στις 21-22 Νοεμβρίου και Ολομέλεια τον Ιανουάριο, 12 Ιανουαρίου. Σημείο 10. Διάφορα δεν υπάρχουν. 11. Προσεχή συνεδρίαση. Το είπα και πριν, καμιά δεκαριά φορές το είπα, ας το ξαναπώ. Η επόμενη μας συνεδρία είναι 21 και 22 Νοεμβρίου. Και 12. Όπως ίσως γνωρίζετε, το απόγευμα γίνεται ακρόαση με θέμα γυναίκες και κλιματολογική αλλαγή. Αν δεν το ξέρετε, οι κλιματολογικές αλλαγές θα έχουν μεγάλ, θα παίξουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας και δυστυχώς δεν θα, το, θα τις υποστούν όλες με τον ίδιο τρόπο στο νότιο ημισφαίριο και ιδίω οι γυναίκες που κατοικούν στο νότιο ημισφαίριο θα τις υποστούν περισσότερο. Αυτά θα με το απόγευμα και ελπίζω να έρθετε πολλές. Κυρίσετε το τέρας τη συνεδρίας.